Όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης, παρακαλώ ας αποχωρήσουν γιατί θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες της Επιτροπής Απασχόλησης στις οποίες ως γνωστό συμμετέχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης. Then we proceed with the voting. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία μόνο μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης. Επιστολή, γνωμοδότηση, υπομορφή επιστολής δηλαδή, σχετικά με αίτηση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θεωρητικές δραστηριότητες Καστίγια ή Λεόν, περιφέρεια της Ισπανίας, ε, υπέρ, όχι, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά ας ψηφίσουμε, παρακαλώ τις κάρτες σας, τα μηχανηματάκια σας και ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά. Have all voted on the... Ψήφισαν όλοι για την επιστολή αυτή. Mr. Becker, you have the chance to vote on... Κύριε Μπέκερ, μπορείτε να ψηφίσετε αν θέλετε. Well, there were 42 votes in... 42 υπέρ, 4 κατά. Επόμενη ε, ψηφοφορία. Πάλι για την επιστολή σχετικά με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάφορες νομικές πράξεις που προβλέπουν τη χρήση κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Ψηφίσουμε λοιπόν επί της επιστολής αυτής. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. ...38 υπέρ, 7 κατά. Και... Περνάμε στον κύριο Μέτσερης... ...και το σχέδιο έκθεσης που έχει συντάξει... We are Θέσπιση κοινού πλησίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Ξεκινούμε με την συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΒΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγγνώμη. Να το ξανακάνουμε λίγο. Συμβαστική BB υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας, συμβαστικής τροπολογίας BB. Πέρας φορές. Εγκρίνεται. Με διαφορά τεσσάρων ψήφων. Συμβαστική C. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. K κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Εποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.47 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 247. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Χίλια συγγνώμη. Έκανα λάθος. Τροπολογία 248 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 250 Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 249. Ωραία, ψηφίστε παρακαλώ τότε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 2.51 ψηφίστε παρακαλώ. The vote is open and the vote is now closed. της Απορρίπτεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική M, μη, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 260, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται παραρτήματα. Page 23. Σελίδα 23. Βλέπετε εκεί την τροπολογία 296. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 298. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 μαζί με την 299 υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Για να το επαληθέσουμε. Ψηφίζουμε επί τις 104 και 299. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία 300 μαζί με την 105. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 300 και την 105. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα της προφορίας. Απορρίπτεται. 106 μαζί με την 301. Πέρα. Τα ποχές μου φαίνεται ότι απορρίφθηκε Απορρίφθηκε λοιπόν 303 υπέρ Τα αποχές εγκρίνεται ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πράγματι. 304 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την τροπολογία 304. Τέλος της ψηφοφορίας. 107. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 120 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Τι υπέρ. Κατά. ποχές εγκρίνεται. U υπέρ. Κατά. ποχές εγκρίνεται. V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα έλεγα αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 132 ψηφίστε σας παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας Α, εγκρίνεται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Με συγχωρείτε. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συμβαστική Y, Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 143. Όχι, όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 15. Μαζί με την 144. Ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 143. Η, καταπίπτει. Συμβαζιστική Z. Z υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 16 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 19, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 20, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αλφα, υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. ΑΒ υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά βοχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά βοχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, όχι, απεσύρθη. Και πάμε στην 158. Υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε επί, ε, του τροποποιημένου σχεδίου έκθεσης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. ψηφίσετε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή. Η εντολή για τη διαπραγμάτευση. Θα ψηφίσουμε και από αυτής. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορία. Ωραία. Ψηφίσαμε και για τη διαπραγματευτική ομάδα. Συγχαρητήρια. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβι... Να ελέγξουμε την τροπολογία 33. Open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτηκε. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε τη 48. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. It's rejected by one vote απορρίπτεται με μία ψήφο συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 όχι 52 συγγνώμη 52 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 52 The is open. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας And it's rejected by Sweden. Απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 56 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ήταν σαν να ψηφίσετε στην 50, για την 54, αλλά δεν ψηφίσετε για την 54. Συμβαστική ήττα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ καταπίπτει Yes, we go to 75. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβι... συμβιβαστική Έλα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την έλλα, τη συμβιβαστική Έλα. Ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 26 ψήφους. Τροπολογία 91. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά. 94 επαναλαμβάνει η πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται συμβιβαστική νη υπέρ κατά να το ξαναδούμε συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική π υπέρ κατά περίπλοκο ε συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη συμβιβαστική πη. Άρχεται ψηφοφορία. And the vote now closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Amendment 100. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 136 υπέρ, με προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές υπέρ, κατά α, να το ξαναπροσπαθήσουμε υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε νομίζω. Για να είμαστε βέβαιοι, την 136 με την προφορική τροπολογία έρχεται ψηφοφορία. πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται με 31 ψήφους. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 139 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 139. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, What happened? If you doing this? it was It was 12.32 if you can accept that. It was 12.32. 12.32 ήταν. Να το ξαναδοκιμάσουμε. Υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Κάτι συνέβη. Κάτι μυστηριώδες. Το δεύτερο τμήμα της 139. Δεύτερο τμήμα της 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα. Ορίστε το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται με 32 ψήφους. Πάμε στην τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 135 Συγγνώμη, 142, όχι 135. Θέλετε τι, θέλετε να τσεκάρουμε, 141. Ωραία, να την τσεκάρουμε. Τσεκάρουμε την 141, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για την 141. απορρίπτεται με 10 ψήφους διαφορά 135 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 καταπίπτει 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 Κάποιος θέλει να τσεκάρουμε την 143 όχι. We check 143 and the 143 τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την 143 και πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με τρεις ψηφούς διαφορά. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 στις αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική C υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 τέλος υπέρ κατά αποχές αποχές ε, εγκρίνεται συγγνώμη ψηφίζουμε από του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ...35 υπέρ, και τέσσερις κατά και τρεις εποχές. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την εισηγήτρια Τάνια Γκοντζάλες Πένιας. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο που έχει να κάνει με τον έλεγχο δαπανών και παρακολούθηση οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων εγγύησης για την ε, νεολαία. Και θα ξεκινήσουμε με την Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να δούμε λοιπόν την 8 να δούμε τι γίνεται εκεί. Έληξε η ψηφοφορία. Άρα λοιπόν είμαστε 28 υπέρ. Sorry. It was a very, it was not a narrow thing. Amendment 9. Περνάμε στην 9 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική K. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά λοιπόν για να τη δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτεται με μία ψήφο παραπάνω κατά 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ την 25 Λίγη. 28 υπέρ λοιπόν. Για την ε, συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη 41 υπέρ κατά αποχές για να δούμε ηλεκτρονικά λοιπόν τι γίνεται με την 41. Άρχεται, πέρας, απορρίπτεται. Πάλι μία ψήφος, η 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για την π, συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Okay. Compromise M, those in favor, those against. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε μετά, αν συμφωνείτε, στην 37 με την προφορική τροπολογία. Εάν όχι, τότε καταπίπτει και αν ναι, θα την ψηφίσουμε με τα όσα προσθέσαμε. Ωραία λοιπόν. Τι θα κάνουμε. Κυρία Σιντάνσκα, έχω αντίρρηση προς την προφορική τροπολογία. Οπότε με τρία μέλη μπορούμε να την μπλοκάρουμε. Ωραία. Μπορείτε να την μπλοκάρετε, οπότε δεν θα ψηφιστεί. Θα περάσουμε λοιπόν. Λοιπόν, η προφορική από τους σοσιαλιστές καταπίπτει. Το ολόκληρο αυτό λοιπόν καταπίπτει. Ξέρετε τι λέει ο κανονισμός. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη που είναι 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να περάσουμε στη συμβαστική Ι, e, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 73 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, α, συγγνώμη, όχι, 92 υπέρ, του Τέρι Ράιντκε, κατά. Να δούμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 92. Άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 106 καταπίπτει και περνάμε στη συμβαφαστική H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 60 καταπίπτει, 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, για το σχέδιο γνωμοδότησης ολόκληρο, Ωραία λοιπόν για το σχέδιο γνωμοδότησης άρχεται η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Υπερψηφίστηκε 36 υπέρ, 4 κατά και 2